Presidente. Non c'è bisogno di microfono. Non Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, ε, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί αν υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Έχουμε στην ημερήσια διάταξη τις δηλώσεις επί Συμβουλίου και Επιτροπής περί SWIFT. Δίνω αμέσως τον λόγο στον κύριο Λόπες Γκαρίγκο που αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Λίστα, τελικά, ο κύριος Υπουργός. Κυρίες και κύριοι, κυρία Επιτρόπε Μάλιστα, τις 24 Τρίτου, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, η Επιτροπή ενέκρινε μία σύσταση προς το Συμβούλιο, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία σύμφωνα με το οποίο θα τεθούν στην ε, διάθεση του Βρήκονου των ΕΥΠΑ κάποια δεδομένα που αφορούν την χρηματοδότηση και τα χρηματοοικονομικά γενικά των τρομοκρατών. Ευθύ αμέσω ενημερώθηκε ο εισηγητή και κάποιοι άλλοι ευρωβουλευτέ, αλλά διαβάστηκε και στο Συμβούλιο. Παραμένουμε πεπισμένοι ότι χρειάζεται να συνάψουμε συμφωνία από αυτό το θέμα και για αυτό συμφωνούμε 100% με τα όσα συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όσον αφορά το πρόγραμμα της ε, παρακολούθησης της χρηματοδότηση των τρομοκρατών. Η Κορεπέρ επίση συζητεί και παρακολουθεί την διεκπαιρέωση της πρόταση και πρόκειται να γίνει και η ψηφορία στο Συμβούλιο των Υπουργών συγκεκριμένα στον αφορά αυτή την σύσταση. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει αυτή την πρόταση και θα λάβουμε υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά και τις απόψεις που σήμερα θα ακουστούν σε αυτό το ημικύκλιο. Συμφωνούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ότι η συμφωνία που θα συναυθεί, η συμφωνία SWIFT θα πρέπει να παρέχει ικανές εγγύησεις. Και συμφωνούμε με την ευαισθησία που δείξατε στο θέμα. Ότι θα πρέπει δηλαδή να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ευρωπαίων. Όπως προβλέπει ο Χάρτης το άρθρο 8, θα πρέπει να γίνει σεβαστή συνθήκη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ε, αυτέ τι βασικέ αρχέ όσον, αφορά τη διαβίωση των προσωπικών δεδομένων, όπω το δικαίωμα τη ενημέρωση, σε σχέση με κάποιο το οποίο τα στοιχεία τα δεδομένα εξετάζονται, όσον αφορά τη διόρθωση επίση για αυτά τα δεδομένα, εάν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αναλυθέ, όσον αφορά την απαλληφή κάποιων εμεί σωστών και θα πρέπει επομένω να ισχύσουν όλα τα σχετικά με την προστασία των δεδομένων χωρί καμία δυσμενή διάκριση. Άρα θα πρέπει ό,τι ισχύει για του πολίτε των ΗΠΑ να ισχύσει και για του πολίτε τη ΕΕ. Θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να συναυθεί μια τέτοια συμφωνία σε σχέση με την διάρκεια της σχετικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ. Ανά πενταετία προβλέπεται. Και όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων τώρα, με τρίτες χώρες, από ό,τι γνωρίζουμε, οι Αμερικανοί έχουν λόγους να θεωρούν ότι υπάρχουν τέτοια δεδομένα που μπορεί να βοηθήσουν τις τρίτες χώρες, ούτως ώστε να μπορέσουν να διώξουν τους τρομοκράτες. Ακριβώς αυτό το οποίο προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Ότι σε τέτοιου είδου περιστάσει, όταν κάποια κρατημένη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν πληροφορίε, έχουν και έχουν πληροφορίε, μπορούν να τι διαβάσουν σε κάποια τρίτα κράτη όσον αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Και αυτό είναι το ζήτημα επομένω τη διαβίβαση των δεδομένων με την ευρεία έννοια και όχι όταν πρόκειται για κάποιον ο φέρεται ω ένοχος, κάποιο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Και επίση τώρα υπάρχουν θέματα τεχνολογικά, υπάρχουν θέματα αποτελεσματικότητα, διότι σε πολλές περιπτώσεις είναι σημαντικό να υπάρχουν πολλά δεδομένα τόσο να μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα την ώρα που θα έρθει η στιγμή της δίωξης του τρομοκράτη των τρομοκρατών. Άπαξ βέβαια και γίνεται αυτού του είδους η των δεδομένων, όσο είναι πιο συγκεκριμένα, με πολύ, πολύ περιχαρακωμένο τρόπο, ούτω ώστε να είναι ο σκοπός η δίωξη των τρομοκρατών. Ακριβώς που είναι η γενεσιουργική αιτία τέτοιου είδους συνθήκων. Γι' αυτό έχουμε τη δεδομένη λεπτομερή αξιόλογη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που παρέχει εγγύσει εγγύσεις τήρηση των ε, θεμελιωτών δικαιωμάτων που λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα αυτή τη συμφωνία που βασίζεται στην αμοιβαιότητα και την αναλογικότητα σε σχέση με τη διαβίωση των δεδομένων και επίση, στον έλεγχο των επιβαλλόμενων ακριβώ όπω έχει προτείνει η Κομισιόν και στον έλεγχο και τον κοινοβουλευτικό που αναπόσπαστα συνδέεται με τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Και έτσι υπάρχουν εγγυήσεις αποτελεσματικότητας αυτής της συμφωνίας. Συμφωνούμε επομένω να προχωρήσει αυτή η πρόταση και ότι θα πρέπει οι επιθυμητέ πληροφορίε να διαβάζονται και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας ενημερώνει στις διαφορετικές φάσεις της διαπραγμάτευσης. Επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση ευκολότερα στα διαβαθμισμένα κομμάτια αυτών των διαπραγματεύσεων, ώστε να μπορεί να τα αξιολογήσει. Και στην δήλωση τη 12ης Δευτέρου του 2010 συμφωνήσαμε να γίνει μια διοργανική συμφωνία με το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και μεγάλη μας χαρά σήμερα σας επιβιώνουμε αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόπες Γκαρίγκο. Το λόγο έχει τώρα η Επίτροπος Σεσίλια Μάλστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, η συλλογή στοιχείων TFTP είναι σημαντική για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία TFTP έχουν βοηθήσει για την ε, πρόληψη ε, τρομοκρατικών επιθέσεων όπω το 2004 στο Heathrow ε, με τις ε, υγρές βόμβες. Επίσης ήρθαμε σε επαφή με τον Υπουργό Ιστορικών ε, Ναπολιτάνο. Γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνει αυτή η συμφωνία, αλλά φυσικά ανησυχούν σε σχέση με το κενό ασφάλειας, αλλά να γίνει αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και να προστατεύονται επαρκώς τα στοιχεία. Ε, τελευταία φορά που συζητήσαμε το θέμα, η Κομισιόν εξέδωσε, ε, μάλλον άρχισε να εργάζεται για μια νέα εντολή, για μια νέα συμφωνία FTP. Η εντολή είναι φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική, εξισορροπεί την διατήρηση της συλλογική μας ασφάλεια, ενώ αντιμετωπίζει τα βασικά δικαιώματα, την προστασία των στοιχείων επί τη βάση του ψηφίσματος του Σεπτεμβρίου πέρσι και του Φεβρουαρίου φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Χένη Πλάσκαρ για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Η Κομισιόν προσπάθησε να συνδεθεί μαζί τη καθώ και με του κοιόδη εισηγητέ για να συντονιστεί μαζί τη και επίση είμαι ευγνώμων στην Προεδρία για τη δουλειά που έκανε προσπαθώντα να περάσει το θέμα από το Συμβούλιο. Προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τι ανησυχίε που εκφράζονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα στοιχεία θα, θα σε επεξεργασία μόνο για στόχου καταπολέμηση τρομοκρατία. Αυτό θα πρέπει να γίνεται ρητά μέσω δικαστική ε, εξουσιοδότηση. Δεν θα δίνονται ε, ε, χίδιν στοιχεία. Τα, τα στοιχεία ΣΕΜΠΑ θα αποκλείονται και επίσης ε, ε, θα διασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν θα ενημερώνει απόλυτα και πλήρως το Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων καθώς και στοχεύουμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία πριν το τέλο του Ιουνίου ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να την ψηφίσει τον Ιούλιο. Για το θέμα των ε, ε, της μεταφοράς ε, μεγάλων όγκων στοιχείων. Ξέρω πως είναι αυτό ανησυχία, αλλά αν δεν υπάρξει αυτό δεν θα υπάρχει και TFTP. Ωστόσο θα διασφαλίσουν οι νομικά δεσμευτικές ε, ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα γίνεται μεταφορά δεδομένων σε μεγάλους όγκους μόνο αν, παρά μόνο αν υπάρχει υποψία. Και η μεταφορά αυτού του στοιχείου θα γίνεται ανώνυμα. Η μεταφορά ε, μεγάλων όγκων στοιχείων είναι ευαίσθητη θέμα και θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε και τον όγκο των δεδομένων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ε, πρέπει ωστόσο να είμαστε ρελεστέ. Δεν θα πρέπει να δούμε πολύ μεγάλη μείωση των όγκων παρά μόνο αυτές τις τα στοχευμένα αιτήματα για μεταφορά ε, στοιχείων. Επίση, ε, θα πρέπει να, γίνονται, να δίνεται ειδική εξουσιοδότηση για να γίνει ε, δίωξη τρομοκράτη σε ευρωπαϊκό έδαφος και αντιστρόφως ανάλογα. Οι Αμερικανοί θα πρέπει να μας επιτρέψουν το ίδιο και η Κομισιόν είναι πρόθυμη να συμμετέχει σε αυτές τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Η εντολή ζητά πενταετή ε, κράτηση στοιχείων για τα, συνολικά, για, για τα στοιχεία αυτά. Είναι το ίδιο με τις χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές και τα σχετικά στοιχεία. Αυτά ισχύουν ε, μέσω της νομοθεσίας περί ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Είμαστε έτοιμοι φυσικά να το συζητήσουμε μαζί σας και να το διαβιβάσουμε τα, τις απόψεις στο Συμβούλιο το τέλος της εβδομάδας. Εγώ πιστεύω πως είναι μια σημαντική βελτίωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνονται υπόψη το, τα αιτήματα των εισηγητών για μια διπλή προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε ε, μια ανταλλαγή FTP, αν και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε εδώ μόνο στην ε, Ένωση, δεν είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων και λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις ε, ισότιμων εταίρων μεταξύ ΙΠΑ και ΕΕ, πράγμα που είναι μακροπρόθεσμος στόχος μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μπουσουτήλ για τρία λεπτά.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 κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο που θα πρέπει να πει το Κοινοβούλιο είναι πως αυτό εδώ το Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία. Φυσικά το Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί συμφωνία ε, με οποιοδήποτε κόστος και φυσικά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και γι' αυτό είναι, αυτό είναι που θα συζητήσουμε σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Μετά από την ψηφοφορία του Φεβρουάριο υπήρχαν δύο σαφή μηνύματα, διδάγματα τα οποία υποκαμίσαμε. Το πρώτο ήταν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νέες αρμοδιότητες, ξεκάθαρες αρμοδιότητες, έχει έχει λόγο και θέλει να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές. Θα το κάνει αυτό επικοδομητικά και υπεύθυνα, αλλά θα ασκήσει τις αρμοδιότητές του. Το δεύτερο δίδαγμα που αποκομίσαμε είναι ότι η πρώτη συμφωνία δεν ήταν αρκετά καλή και χρειαζόταν ε, βελτίωση. Εγώ καλωσορίζω την ε, ταχύτητα της Κομισιόν και την ετοιμότητά της ε, μας ε, έδωσε μια νέα εντολή τόσο σύντομα. Ε, επίσης προσβλέπω στην έγκριση αυτής της εντολής εξίσου σύντομα από το Συμβούλιο των Υπουργών. Όπως είπα το Ευρωκοινοβούλιο επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία και έχουμε ε, τοποθετήσει τις λεπτομέρειες των όσων θα επιθυμούσαμε στο ψήφισμα το οποίο βρήκε ευρεία συνένεση εδώ στο σώμα και σίγουρα βρήκε τη συνένεση των μεγαλύτερων ομάδων. Τώρα, ε, μεγάλη όγκη στοιχείων ε, χίδιν είναι ένα σημαντικό θέμα για μας και ξέρετε ότι αυτό που επιθυμούμε θα απαιτήσει ένα εκ νέου προβληματισμό και όχι μόνο από πλευρά των εταίρων μας τη ΕΠΑ αλλά και από δική μας πλευρά. Τι ακριβώς θέλουμε δηλαδή εδώ στην Ευρώπη για εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να έχουμε τα το δικό μας ευρωπαϊκό TFTP και πώς θα το καταφέρουμε αυτό, αλλά σαφώς τα hidden στοιχεία είναι ζήτημα και είναι ζήτημα που δεν, μπορεί να το, δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις λεπτομέρειες όταν θα συζητήσουμε με τους ε, τέρους μας στο Κογκρέσο στις ΕΕΠΑ όταν θα μεταβεί εκεί μια αποστολή του Κοινοβουλίου Νομίζω πως έχω τρία λεπτά, Πρόεδρε, γι' αυτό και θα συνεχίσω για 30 ακόμα δευτερόλεπτα, μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν την επόμενη εβδομάδα που θα μεταβεί η αποστολή του Κοινοβουλίου στις ΕΙΠΑ θα συζητήσει το θέμα με τους ε, ομολόγους του αλλά και με τις αρχές των ΗΠΑ και αυτό θα φροντίσουμε ώστε να γίνει με επικοδομητικό τρόπο. Θέλουμε να πάμε εκεί για να δείξουμε στις Αμερικανικές αρχές ότι το εννοούμε, ότι επιθυμούμε τη συμφωνία, αλλά και ότι και εμείς έχουμε ανησυχίες και θέλουμε αυτές οι ανησυχίες να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Και ακόμη μια φορά ζητώ συγγνώμη που σας διέκοψα, αν έκανα λάθος. Είχα διαβάσει δύο λεπτά αντί για τρία. Και τώρα έχει το λόγο η κυρία Μπερτζίτ Σίπελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαφωνήσω σε ένα σημείο με τον προλαλήσαντα. Το δικό μου συμφέρον δεν είναι να έχουμε το ταχύτερο δυνατό συμφωνία, αλλά το καλύτερο δυνατό συμφωνία ή την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Η ποιότητα προέχει τη ταχύτητα. Ε, θα ήθελα να κάνω και μια άλλη εισαγωγική παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ήδη έχει απορρίψει μια συμφωνία. Και πέρα από του πολλού λόγου ουσία, υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο που ήταν η μη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή την εβδομάδα ε, για λόγους εκτάκτους και επίκαιρους αποφασίσαμε να μην λάβουμε καμία απόφαση στο Κοινοβούλιο και είπαμε και το Συμβούλιο να αναβάλει τις αποφάσεις του μέχρι να έχουμε εμείς τη δυνατότητα να αποφασίζουμε. Με εκπλήσει λίγο που υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δεν παίρνουν σοβαρά τις ίδιες μας τις αποφάσεις και θεωρούν ότι καλά δεν πειράζει, ας αποφασίσει το Συμβούλιο. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια μεταχείριση στις ίδιες μας τις αποφάσεις. Εγώ επιμένω και το Συμβούλιο να αναβάλει την απόφαση του μετά την 6η Μαΐου όταν θα έχουμε αποφασίσει εμείς. Και είμαι βέβαια βέβαια ότι δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία και έχουν και κατανόηση για αυτό που συμβαίνει. Τώρα, έχουμε ε, στο σχέδιο αυτό καθ' αυτό της εντολής. Καταλαβαίνω και κατανοώ αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει να ανταποκριθεί στα δικά μας λύματα, αλλά χρειάζεται μεγάλη αλλαγή η εντολή αυτή. Αν θέλετε κατά πλειοψηφία να συμφωνήσει το κοινοβούλιο μας, γιατί η σημερινή εντολή δεν προσφέρεται και δεν είναι αρκετά φιλόδοξη ως προς αυτό το στόχο. Η μαζική μεταφορά δεδομένων είναι ένα πρόβλημα που παραμένει ανεπίλητο. Μας λένε οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πρόκειται για 5 με 10 πρόσωπα ε, συγκεκριμένα κάθε μήνα. Γιατί να στέλνουμε εκατομμύρια πληροφορίες για Διάφορου πολίτε τη Ένωση. Είναι τελείως δυσανάλογα αυτά τα πράγματα. Και θέλω να πω και πάλι στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Ε, υποτίθεται ότι είναι υπαρξιακή σημασία σε αυτή η συμφωνία ε, ω επιπλέον μέτρο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό δεν το καταλαβαίνω ούτε είναι αρκετά τεκμηριωμένο. Παραμένει προβληματική και η περίοδος στήριση των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οθήκευσή του και αυτό δεν το λύνει η εντολή. Χρειαζόμαστε μια δικαστική αρχή σε ευρωπαϊκό έδαφος που να μην ελέγχει μόνο την αίτηση των ΗΠΑ ως πρωτοπαραδεκτό αλλά και τα στοιχεία ε, και την ε, εξέβρεσή τους όπου και αν συμβαίνει αυτή. Επίσης θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες που διέπουν τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη ε, συμφωνία και φιλόδοξη εντολή για να ε, έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προστασία των δεδομένων των πολιτών. Και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς σκέφτεστε να εξασφαλίσετε ότι θα διαβάζονται μόνο τα συγκεκριμένα στοιχεία που ζητούν. Πώς θα γίνει αυτό και πού θα γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού. Έχετε και άλλες προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζίπελ και τώρα για τρία λεπτά έχει το λόγο η κυρία Ένες Πλάσκερτ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να καλωσορίσω τη σημερινή συζήτηση όπου το Κοινοβούλιο εκθέτει τις δικές του προσδοκίες σε σχέση με τις ε, ε, διαπραγματεύσεις. Ε, το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει αυτή την εβδομάδα για το ψήφισμά του είναι ατυχές, αλλά αυτό θα πρέπει να εμποδίσει το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει το, ε, την πρόταση όπως έχει προγραμματιστεί. Είναι πολύ σημαντικό και όλοι γνωρίζουν την πρόταση ψηφίσματος. μπορώ μόνο να πω ότι εκτιμώ το νέο πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν τόσο το Συμβούλιο όσο και η Κομισιόν για συνεργασία δηλαδή με το Ευρωκοινοβούλιο. Για την, οδηγία, την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων, εμείς θέλουμε να διαπραγματευτούμε ίσα δικαιώματα ασχετά με την εθνικότητα του ατόμου που, του οποίου τα στοιχεία μεταφέρονται. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, για παράδειγμα, όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση, την διαγραφή, την αποζημίωση και την ε, και εδώ θα ήθελα να με ενημερώσετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Και έπειτα η αρχή της αναλογικότητας είναι μια ανάγκη αδύρυτη για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας. Και το γεγονός ότι οι πάροχοι στοιχείων δεν είναι σε θέση να αναζητήσουν ένα συγκεκριμένο μόνο πρόσωπο με ξεπερνά και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει τα η μαζική μεταφορά στοιχείων να ε, προσεχθεί. Εγώ έχω αφιβολίες για το αν θα λυθεί αυτό το θέμα επί τη βάση της, ε, των οδηγιών που υπάρχουν για τις ε, διαπραγματεύσεις. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η αμοιβαία νομική αρρωγή δεν είναι η κατάλληλη βάση για την αίτηση στοιχείων με βάση το TFDP. Εξάλλου αυτό δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει για τις μεταφορές ανάμεσα σε τρίτες χώρες, αλλά απαιτεί προηγούμενο εντοπισμό ε, των στοιχείων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι διαπραγματεύσει να εστιαστούν στην εξέβρεση μια λύση ώστε να είναι συμβατά όλα αυτά. Φυσικά θα μπορούσαμε να επιμείνουμε για το νέο σχεδισμό του TFTB, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν εξαρτάται από εμά και γι' αυτό μπορώ μόνο να παρατρύνω το Συμβούλιο και την Κομισιόν να, ε, όπως και ο κύριος Μπουσουτήλ, για να ε, υιοθετήσουν την απόφαση αυτή αμέσως. Θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να ε, εισηχθεί μια ευρωπαϊκή λύση νομικά βάσιμη, νομικά στριγμένη για τη μεταφορά των στοιχείων. Η αποθήκευση, η μεταφορά μάλλον και αποθήκευση στοιχείων από μια ξένη δύναμη, ακόμα και είναι αυτή ο καλύτερος μας φίλος, είναι δυσανάλογο ε, ζήτημα, σημαίνει μεγάλη απόκληση από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την πρακτική. Το κράτο δικαίου είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα στο να αξιολογήσει μια προτινόμενη συμφωνία όπως αυτή εδώ. Γι' αυτό και θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μπορούμε να ενεργούμε ισότιμα Ω ισότιμο εταίρο με τη ΣΥΠΑ. Μπορώ, θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω ακόμη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ορίσει τι αρχέ επί των οποίων θα συνεργαστεί με τρίτου ε, ε, ε, εταίρου συμπεριλαμβανομένε τη επιβολή του δικαίου. Η νόμιμη κατεργασία προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη και τώρα το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει όλα αυτά να τα θέσουν σε απόλυτη εφαρμογή και να διαπραγματευτούν συμφωνίες που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τόσο της Ένωσης όσο και των ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Γιάνν Άλμπρεχτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Προεδρία και την Επίτροπο κυρία Μάλμστρομ για τις παρατηρήσεις της. Η Προεδρία έχει δίκιο. Στη συμφωνία TFTP πρόκειται για συγκεκριμένες αρχές, για αρχές συνταγματικές και θεμελιώδεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, άρθρο 8 του χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 8 της ΕΣΔΑ της ευρωπαϊκή σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας δικαίου, άρθρο 6 και άρθρο 13 για σωστές διαδικασίες και αναλογικότητα ουσιαστική και πραγματική με τη συνταγματική έννοια, έτσι, την έννοια του συνταγματικού δικαίου και το τονίζω. Δεν είναι να έχουμε απλώς μία αίσθηση αναλογικότητας. Όχι, τεκμήρια, συγκεκριμένα στοιχεία για την αναγκαιότητα, γιατί είναι σκόπιμο ένα μέτρο και ποια είναι ακριβώς ε, ωφέλεια που θα έχουμε. Και θα ήθελα να τονίσω το εξή. Ορισμένοι εμπειρογνώμονε αλλά και ιδιοκτικέ αργέ έχουν πει επανειλημμένα ότι η μαζική ε, διαβίβαση ε, δεδομένων χωρίς την παραμικρή υποψία δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι είναι παραγωγική. Δεν αρκεί από ε, η μεταβίβαση και μόνη ε, για να ε, δώσει τα στοιχεία που χρειάζονται. Αν δεν έχουμε συγκεκριμένες υποψίες, δεν μπορεί κανείς ε, να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποτρέψουμε τη μαζική διαβίβαση δεδομένων. Αλλιώς αυτό θα ήταν παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των διεθνών συμβάσεων και αυτό μέχρι τώρα έχουν αποφανθεί τα περισσότερα δικαστήρια στην Ευρώπη και το Μάρτιο το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας, ξέρετε. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να ε, απεμπολίσει τις θέσεις που υποστήριζε μέχρι τώρα. Αλλά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και μετά τις διαπραγματεύσεις να είναι ε, βέβαιο ότι διαφυλάσσει την νομιμότητα και ενδεχομένω να επιφυλαχθεί να προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη συνέχεια. Παρακαλώ λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ε, υποστηρίξει ενώπιον των Ηνωμένων Πολιτειών τη θέση του Κοινοβουλίου και να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Αλλιώ δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει. Ο κύριος Στάνοκ για δυόμιση λεπτά. την ερική Συμφωνία για το Συμβημί είπα. την υποστήριξη πολιτική ομάδα όσον αφορά την παρακολούθηση και ανείχνευση των ε, τρομοκρατών όσον αφορά αυτά τα οικονομικά δεδομένα, φυσικά με την επιλέξη κάποιων ε, ρητρών ασφαλεία. Ε, και βέβαια δεν είπαμε με τίποτα να υπάρχει ούτε μηχανισμό ούτε δουλειότητα γιατί οι Αμερικανοί αποτελούν μια εγγύηση για τα δικαιώματα όλων. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερο, όχι λιγότερα και να παραμείνουν στην πρωτοπορία ε, την αντιτρομοκρατική. Εμεί θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το SWIFT, ούτω ώστε να μπορέσουμε να φημώσουμε οικονομικά την ε, τρομοκρατία και να προσθέσουμε και πιο στον ελληνικό τον κόσμο. Όμω ήταν θλιβερή η καταψήφιση, παρόλο το ότι δεν με εξέπληξε, διότι αναμφίβολα το ε, Κοινοβούλιο κοιτούσε την ισορροπία δυνάμεων και ήθελε να δείξει το ότι είναι πιο δυνατό με την στιγμή τη Λισαβόνα. Όμως Έχουμε την νέα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Επομένως, ουδέν κακόν, αμυγέ καλού. Και έτσι ίσως αυτό να είναι ξυπνητήρι για την κυβέρνηση Ομπάμα. Μια που αντίθετα με τους προκατόχους ε, δεν έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται, τι, κάνει, τι, τι, τι, τι ρόλο παίζουν τα θεσμικά όργανα και ιδίω το, το Κογκρέσο, το Κοινοβούλιο και δεν κάθεται να, να, να ακούσει τους διπλωμάτες, τους ε, γιατί θυμάστε ο κύριος Μπούζεκ με τον κύριο Κλίνο και τους συμβούλους του πόσο εύστοχα τα είχαν συνοηθεί και επομένω να, τα αγνοούμε όλα αυτά, αυτό είναι αφελές αλλά και υπερφύαλο. Η ΕΠΑ έχουν άλλωστε εδώ στο Κοινοβούλιο ένα λόμπι, αόρατο αλλά πολύ δυνατό. Ε, Ταϊβάν, Κολομπία, Ισραήλ, Κίνα, Ινδία, αυτοί επενδύουν πάρα πολλά για δημόσιες σχέσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Οπότε και με διπλωματικούς ελιγμούς θα πάνε καλά. Όμως, είπα, ενώ έχουν τεράστιες δυνατότητες δεν τις εκμεταλλεύονται. Έχουμε τη διμερή αντιπροσωπεία στο, στο Βέλγιο που είναι η διπλάσια από την αντιπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βίλιαμ Κέναρτ, πάντως, ο επικεφαλής, ε, μας εκτιμά εμάς και το έργο μας και αυτά νομίζω διαβάζονται όπως πρέπει στην Washington. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις μας ε, με, την Αμερικανική κυβέρνηση και, με, και ο κύριος Μπάιντεν επίσης είναι πάρα πολύ καλό θετικό στοιχείο γιατί φυσικά το, αυτό που θέλω προς το πω είναι να τα πάμε καλά. Επομένως, να πάει πάρα πολύ καλά το SWIFT και όσον αφορά τα δεδομένα των υπηρετών, το PNR, ε, χωρίς η συζήτηση να περιέχει αντιφάσεις να διφορούμε. Ε, ο ε, η κυρία Ευχαριστώ. Κυρία Βερζιά, κύριε Πρόεδρε, αν δεν σας πειράζει. Ε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά συζητούμε για την εντολή Συμβουλίου και Επιτροπής για το σχέδιο SWIFT. Το σχέδιο εντολής που σήμερα μας ε, υποβάλλεται ε, υιοθετεί βεβαίως ένα τμήμα των αιτήσεων του ε, Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2009 από το τότε ψήφισμα αλλά παραμένει ε, η κατάσταση προβληματική όπως είναι ο χρόνος στήριξη των δεδομένων η δυνατότητα προσφυγής των πολιτών η νομοθεσία στις ΗΠΑ είναι αρνητική εισάγει διακρίσει κατά των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτών τρίτων χωρών εκτό των ΗΠΑ. Αυτό το αναγνωρίζουν ακόμα και οι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τεράστιο πρόβλημα επίση ω προ την αναλογικότητα, την δυσανάλογη κατάσταση αυτή. Και εσεί η ίδια, κυρία Επίτροπε, μα είπατε ότι παραμένουν ανησυχίε σε αυτέ τι μαζικέ μεταφορέ μεικτών δεδομένων. Λυπάμαι σε ό,τι με αφορά εγώ δεν εμπιστεύομαι τη λειτουργία των Αμερικανικών αρχών η θεωρία της υποψίας δεν μπορεί να είναι ικανοποιητική. Γνωρίζουμε οι Αμερικανοί τι ε, ζημίες έχουν προκαλέσει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όπως είπε η κυρία Σίπελ, η ε, ποιότητα προέχει της ποσότητας. Βεβαίως να υπάρχει ε, δυνατότητα πραγματικού ελέγχου στα στοιχεία που διαβιβάζονται. Χρειαζόμαστε ακόμα εγγυήσεις για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας, των συμπολιτών μας και όσων ζουν στην Ευρώπη, ανδρών και γυναικών. Ήδη χαιρόμαστε για τις πρόοδους που έχουν γίνει, αλλά είναι ανεπαρκείς, επαναλαμβάνω. Οι πολίτες μας έχουν δικαίωμα ε, στην ασφάλεια, αλλά παντού. Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει προστασία της ιδιωτικής ζωής, αλλά ε, είμαστε υποχρεωμένοι να σας προειδοποιούμε και να ε, ακούμε τη συνείδησή μας η αρχή της αναλογικότητας ε, δεν γίνεται πάντα σεβαστή. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κυρία Βέρτζατ, εγώ ήθελα να διευκρινίσω μόνο, γνωρίζω πολύ καλά ότι είστε κυρία, αλλά στα Ιταλικά ο όρος ονορεύολε είναι το, σημαίνει τόσο κυρία όσο και κύριος. Αξιότιμος ή αξιότιμη. Γι' αυτό είπα και ονορεύολε Βερζάτ. Δεν υπήρχε ε, καμία κακή πρόθεση. Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω την εγκυρότητα της διευκρινήσής σας και την ανάγκη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην, χάνει την, να μην ξεχνά το ρόλο και τη σημασία και τη χρήση της Ιταλικής γλώσσας που τόσο έχει προσφέρει στην, Ιταλική, στην Ευρωπαϊκή συγγνώμη, κουλτούρα. Έρχομαι στην συζήτηση και ήθελα να πω ότι μετά από το αστιάκι αυτό που έγινε εκείνη μάλλον την έκδοση του κειμένου το οποίο απορρίφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε βέβαια να δώσουμε τον επίγοντα χαρακτήρα και ε, του θέματος να μην αποδυναμώσουμε με κανένα τρόπο ένα, μια σημαντική απέτηση της Ευρώπης να υπεραμεινθούμε ε, ε αυτών εναντί της τρομοκρατίας. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, μια αναλογικότητα. Αυτά δεν θα πρέπει να θυσιαστούν στο, τα δικαιώματα των, ε, των πολιτών, τα δικαιώματα της ιδιωτικής, στην ιδιωτική ζωή. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι εγγυημένα, όπως είναι εγγυημένα από αυτή τη νέα διατύπωση της της Κομισιόν που δέχτηκε όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο, τη δυνατότητα οι πολίτες να μπορούν τόσο σε διοικητικό και έδρα όσο και σε νομική έδρα, δικαστική μάλλον έδρα, να μπορέσουν να αμφισβητήσουν διάφορες, ε, διάφορα θέματα με βάση το σύστημα SWIFT. Οι βελτιώσεις λοιπόν θα πρέπει να θεωρήσουμε πως είναι σωστές αυτές τις οποίες επέφερε η Κομισιόν και θα πρέπει να σκεφτούμε πως είναι απαραίτητη συνεργασία με τις αρχές των ΗΠΑ στο θέμα των οικονομικών συναλλαγών ώστε να μπορέσουμε όντως ε, να κάνουμε πρόληψη όσον αφορά την ε, τρομοκρατική απειλή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και η Ευρώπη πρέπει να θυμάται πως πρέπει να ε, αμυνθεί έναντι της τρομοκρατίας. Είχαμε πάρα πολύ σημαντικές αποδείξεις, εξαιρετικά σοβαρές και να διασφαλίσουμε επίσης και τη δημοκρατική ροή των ε, στοιχείων ε, την οποία θα επιβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή πιο σοβαρή προστασία που θα μπορούσε να γίνει για τα προσωπικά στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών και την προστασία των δικαιωμάτων τους που θα πρέπει να υποστηριχτεί σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε βήμα. Πολλές υποδείξεις δώσαμε εμείς οι Ευρωβουλευτές και αυτό ε, λέει πολλά όσον αφορά τον νέο ρόλο, τον ενδυναμωμένο ρόλο του Κοινοβουλίου με βάση τη Συνδική. Εξάλλου, συμφωνία προβλέπει αμοιβαιότητα από πλευρά των ΗΠΑ. Αν δηλαδή η Ευρώπη φτιάξει ένα τέτοιο ε, σύστημα ελέγχου των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, κατά της τρομοκρατίας θα πρέπει να κάνει το ίδιο. Θα πρέπει να μπορέσει η ίδια να έχει εισρωή. Το σύστημα PNR θα το συζητήσουμε αργότερα και ισχύουν ναι, ίδια, τα ίδια επιχειρήματα Πρόκειται για την αναγνώριση των ε, επιβατών πάντοτε με στόχο την καταπολέμηση τρομοκρατία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Μποργέτζιο, Το λόγο έχει ο κύριο Τράσερ για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Εμείς από το Βαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλουμε συμφωνία και θέλουμε να έχουμε καλύτερη σχέση με τους Αμερικανούς μας φίλους παντού, κυρίως όμως ε, στην ασφάλεια. Θέλουμε και καλή συμφωνία και ε, γοργή συμφωνία. Και τώρα πραγματικά πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι η στιγμή που αντικατοπτρίζει και το πνεύμα της ε, Λισαβόνας. Όσο σπάνια στο παρελθόν. Μετά το ψήφισμα που, πήρε το, ε, που ενέκρινε το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβρη, ε, το Συμβούλιο στα τέλη του έτους. Ε, στη συνέχεια ακολούθησαν συζητήσεις τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και στο Κοινοβούλιο και τώρα έχουμε μια κατάσταση που είναι καλό παράδειγμα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά κυρία Επίτροπε και σας και το Συμβούλιο για αυτή τη νέα κίνηση, τη νέα αρχή και εσείς και η κυρία Ρέντιν κυρίως και αυτό ε, είναι ένα παράδειγμα αποτελεσματικότητας που θέλει να βλέπει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι από κοινού καταλήγουμε σε λύσεις. Και όχι μόνο ο Ευρωπαίος πολίτης, αλλά το βλέπουν όλοι εκείνοι που είναι σήμερα παρόντες. Και θα ήθελα να ε, απευθυνθώ στους φίλους από το Ρήνο, από την Αυστρία και όλες τις ομάδες επισκεπτών που παρευρίσκονται σήμερα στο ημικύκλιο. Κυρίες και κύριοι, εμείς δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα. Αγωνιζόμαστε για τις λύσεις τους. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε βρει πολύ καλές ε, ε, αφετηρίες ε, για λύσεις, είτε πρόκειται για το θέμα της μαζικής μεταφοράς στοιχείων, για τις τρίτες χώρες, για τη διάρκεια ε, διατήρηση των στοιχείων για την προσφυγή στα δικαστήρια αυτά και τώρα θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και εκπλήσουμε λίγο από τους συναδέλφους των Πρασίνων και της Ενωτικής Αριστεράς που τότε δεν είχαν υπερψηφίσει το ψήφισμα αρνήθηκαν να συνεισφέρουν και τώρα έρχονται και επικαλούν να τηρηθεί το ψήφισμα επικαλούνται ε, Μα ελάτε κι εσείς ξανά πίσω στην κοινή προσπάθεια για να διαπραγματευτούμε μαζί για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι καλή η προσπάθεια και έτσι θα πρέπει να δουλεύουμε στο μέλλον. Το είπατε άλλωστε και εσείς στη δηλώση σας. Εκεί θα οικοδομήσουμε το TFTP βεβαίως και θα το επιβάλλουμε, θα χρειαστούμε αυτό το εργαλείο και επίσης το χρονοδιάγραμμα να το τηρήσουμε όπως ε, το είχατε σκεφτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα πριν τις ενές διακοπές να ε, συζητούμε για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και ελπίζω να τα ε, εγκρίνουμε κιόλας. Για να τελειώνω, θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνετε εσείς τις διαπραγματεύσεις ε, αντικατοπτρίζεται και στο πρόγραμμα δράσης και μπορεί και εκεί να βρει συνέχεια. Για τη συμφωνία για το PNR, το ΣΥΣ και διάφορα άλλα ε, συναφή. Ευχαριστώ. Grazie onorevole Strasser. La parola ora per 2 minuti e 30 all'onorevole Kinga Gons. Ευχαριστώ κυρία Kinga Gons για 2,5 λεπτά. Köszönöm Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε να σας υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν είχαμε κάποιες αρνητικές εμπειρίες. Θυμάστε και την αρνητική ψηφορία. Όμως από τότε τα πράγματα πήραν καλύτερο δρόμο. Η σημερινή συμφωνία είναι πολύ πιο καλή από ότι η προηγούμενη και ελπίζω να συναυθεί αυτή η συμφωνία οριστικά, να ολοκληρωθεί πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα είναι πολύ πιο ανοιχτή στι τάσεις τους οι Αμερικανοί. Σύμφωνα σε αυτές τις έξι επιμέρους προτάσεις, πιο εύκολα από ό,τι το παρελθόν. Καλύτερο συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων, καλύτερη συνεργασία υπάρχει. Πολύ θετικά όλα αυτά. Ακόμα και το ότι είναι εδώ η κυρία Σεσίλια Μάστρομ παρίσταται εδώ και έρχεται στην Επιτροπή μα και μα ενημερώνει τακτικά συνοείται με την Επιτροπή, συνοείται ε, με τους συζητητές. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας για το μέλλον. Ούτως ώστε να έχουμε και άλλες αξιόλογες συμφωνίες στο μέλλον. Ποια είναι τα επόμενα βήματά μας. Τονίζω και αυτό το οποίο είπαν και άλλοι. Έχουμε δεσμευτεί. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ότι πρέπει να με τέτοια συμφωνία και σύντομα μάλιστα να είναι συμφωνία καλή, αξιόλογη, να καλύπτει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Να λαμβάνει πρόσθετη προστασία των δεδομένων, θέλουμε να υπάρχει συνυπευθυνότητα φυσικά για να καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες. Φυσικά ξέρουμε ότι είναι μια ολόκληρη εξίσωση κατά της τρομοκρατίας και είναι μόνο μια μεταβλητή η ανταλλαγή των ε, δεδομένων. Έχουμε αυτή την εντολή, έχουμε ένα σωρό στοιχεία, κάποια ερωτήματα απαντήθηκαν, κάποια όχι. Πριν από λίγο αναφέρθηκαν τέτοια ερωτήματα, τα οποία ακόμα πρέπει να συζητηθούν και να ξεκαθαριστούν. Έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα δεκαπενθήμερο λόγω των, των διαταραχών στην κυκλοφορία πήραμε τώρα αυτή την παράταση που είναι θετικό γιατί μέχρι να ψηφίσουμε θα τα έχουμε σκεφτεί ξανά. Να έχουμε αυτά τα έξι σημεία που ακόμα δεν έχουν επιληθεί οι επιφυλάξει, οι ερωτήσει του Κοινοβουλίου. Ελπίζω. Σε επόμενο δεκαπενθήμερο θα δοθούν κάποιες απαντήσεις και το Συμβούλιο δεν θα απαντήσει πριν εμείς έχουμε καταλήξει κάπου. Ευχαριστώ κυρία Κίνγκα Γκόνς και τώρα. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Λούντφορτ. Να χαιρετήσω και εγώ τους ε, παρόντες ακροτές καθώς και όσους μας παρακολουθούν στο ίντερνετ. Φαίνεται πως είναι πολύ άριθμοι. Οι εργασίε μα έχουν πολλού ακροατέ λοιπόν μέσω των νέων τεχνολογιών και αυτό μα χαροποιεί ιδιαίτερα. Η κυρία Λούτφορντ. Η Κομισιόν σαφώς και άκουσε το σχέδιο εντολή είναι μια μεγάλη βελτίωση των προηγούμενων ε, εντολών. Οι συνάδελφοι υπογράμμισαν τις ανησυχίες που παραμένουν, δεν θα τις επαναλάβουν. Να ευχαριστήσω την κυρία Χένης Πλάσκαρτα για τη δική της σκληρή δουλειά από πλευρά του Κοινοβουλίου. Και να πω και κάτι για το πλαίσιο. Η πρόσφατη πρόοδος αποτελεί τιμή στο τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι εταίροι συμπεριφέρονται μεταξύ τους με σεβασμό και ακούν οι μεν τους δε. Κομισιόν πιστεύω πως, ε, εκτός από την Κομισιόν, πιστεύω πως και οι αρχές των ΗΠΑ έχουν κάνει αυτή την προσπάθεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη Κνάρτ ως προς αυτό γιατί έχει λάβει υπόψη του τις εργασίες του Κοινοβουλίου, ίσως πολύ περισσότερο από ότι ορισμένα κράτη-μέλη της Ένωσης. Τώρα χρειάζεται το Συμβούλιο να κάνει την ίδια προσπάθεια και να υιοθετήσει την ε, προοδευτική αυτή εντολή. Το Συμβούλιο την περασμένη φορά δεν μπόρεσε να έρθει να μας ρωτήσει εγκαίρος ώστε να φτιάξουμε την διάμεση συμφωνία. Τελευταία δεκαετία και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Οι αρχές ε, των ΗΠΑ και της Ένωσης έχουν αντιδράσει με κοινό και συντονισμένο τρόπο για να αντιμετωπίσουν ε, τρομοκρατικές ε, απειλές και πολλές φορές οι κυβερνήσεις πολλές φορές έχουν δεχτεί κατηγορίες για το πώς έχουν αντιδράσει. Δεν θα πρέπει πια όμως να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει οι βασικές μας αρχές για την αναλογικότητα να ισχύσουν, να ελέγξουμε τα σχέδια ε, με σωστό τρόπο και από ό,τι κατάλαβα η Επίτροπος μάλιστα ακριβώς αυτό προεκτήθεται να κάνει ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα για τα κενά, την επικάλυψη και τα επικαλυπτόμενα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα χωρίς να ε, θίξουμε τις ελευθερίες μας. Ευχαριστούμε κυρία Λούτφερ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σαρτζεντίνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είτε έχουμε ψήφισμα είτε όχι. Την περασμένη φορά το Συμβούλιο μας άκουσε πάρα πολύ καλά και ξέρει τι του αναλογεί και τι πρέπει να κάνει. Το Κοινοβούλιο ανησυχεί για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και την προστασία των δεδομένων τους. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Και με θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορεί κανείς να κάνει μια απλή ανάλυση κόστους ωφέλους και τελείως υπόθεση. Και τι είναι αυτά ε, με τη μαζική μεταφορά των δεδομένων, γιατί δεν μπορούν τεχνικά λέει, ε, έχουν την κατάλληλη επεξεργαστή. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω καταρχήν και ε, θεωρώ ότι μάλλον το θέμα είναι κόστους και οικονομίας και σας είπα προηγουμένως, όταν ε, το θέμα τα θεμέλια δικαιώματα δεν μας απασχολεί το πόσο κοστίζει η όλη υπόθεση. Και το Κοινοβούλιο ε, λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να είναι ισότιμο εταίρο στη διαπραγμάτευση και να μην περιμένει να του στέλνουν ΟΠΑ πολιτείε όταν δεήσουν κάποια αντίγραφα ή ορισμένες προφορίες. Εμείς περιμένουμε να παίξετε σοβαρά αυτό το ρόλο. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο και να σα ζητήσω να λάβετε υπόψη σας ε, τη ε, συνθήκη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την ΕΣΔΑ, που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ε, της εντολής σας και θα πρέπει να είναι και στο αποτέλεσμα των όσων πετύχετε. Ελπίζω να κάνετε καλή χρήση την εντολή που σας δίνουμε και σας δώσαμε και την περασμένη φορά. Καλή χρήση της εντολής αυτής και θα περιμένω να δω το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη. Το λόγο τώρα έχει. Ο κύριος Μάρεκ Μιγκάλσκι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, σήμερα η ΕΠΑ είναι η πρώτη υπερδύναμη στον κόσμο, οικονομική και στρατιωτική. Είναι προς μεγάλη μας τύχη που είναι σύμμαχος και φίλος και συμμερίζεται τις ίδιες αξίες και αρχές. Θα πρέπει αυτό να το τιμούμε, θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις είπα όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επί δεκαετίες υπεραμείνεται της Ευρώπης κατά του Κομμουνισμό. Ε, σήμερα έχουν κλείσει 40 χρόνια από την απελευθέρωση από τον κομμουνισμό τη Ανατολική Ευρώπη. Υποστήριξε πάντοτε, είπα, τον ελεύθερο κόσμο. Δηλαδή, τώρα θέλει να παραστατεύσει τον ε, ελεύθερο κόσμο να παραμείνει ελεύθερο από την τρομοκρατία. Τεχνολογία, πόροι χρειάζονται και εκεί και εδώ. Και θα ήταν ντροπή να μην μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Να λοιπόν, τι νόημα έχει αυτή η συμφωνία. Να βοηθήσουμε τη ΣΥΠΑ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Καμία αμφιβολία περί τούτου. Φυσικά και θα πρέπει να περισσώσουμε και προστατεύσουμε τις αξίες που μας διέπουν, αλλά Κομισιόν και Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάτσουν και να βρουν λύσεις να τα διεκπαιρεώσουν όλα αυτά. Επομένω, σήμερα αυτό διατρανώσουν την πολιτική μα βούληση να υπάρξει αυτή η συμφωνία και αυτό θέλουμε να γίνει. Η ΔΕ είπα θα πρέπει να κάτσουν και τα βρούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε φίλοι. Και ακριβώ η αρχή τη εταιρική σχέση πρέπει να διέπει τι σχέσει μα. Και τώρα, Σφένσον. Ε, η κυρία Σβένσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που είχε σημειωθεί. Παρά όλε τι δεξιότητε. Από τότε που είπαμε ότι απορρίπτουμε το σχέδιο τη σχετική συνθήκη. Διατυπώσαμε κάποια αιτήματα, κάποιε προτάσει και είπαμε ότι αν είναι έξυπνη το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να κάτσουν να ακούσουν ποιε ήταν οι επιφυλάξει μα το Φεβρουάριο και να ανταποκριθούν αναλόγω. Διότι Ζητήσαμε προστασία τη ελευθερία και των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων. Είπαμε ότι αυτή είναι η βάση. Για να υπάρχει κράτο δικαίου. Και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν τώρα να θέλουμε να υπάρχει τέτοιου είδου χίδιν μαζική διαβίωση δεδομένων. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί αν θέλουμε τέτοιου είδου μαζική διαβίωση δεδομένων, τότε ανακατεύονται τα ξερά με τα χλωρά και καίγονται. Δηλαδή με του φέρουμε ω ύποπτου οι αθώοι. Επομένω, θέλουμε όταν υπάρχουν βάσιμε υποψίε, τότε να επιτρέπει διαβίωση των δεδομένων. Πάντα για κάποιο φυσικό πρόσωπο. Τώρα, να δούμε την πολιτική πλευρά του ζητήματο. Τι θέλουμε να δούμε. Τα μέτρα που θα πάρουμε να δίνουν το βάρος τους στην στη, στη τεχνολογική πλευρά ή στο θέμα της ε, ε, ε των δικαιωμάτων. Για μένα είναι προφανής η απάντηση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ένα λεπτό ο κύριος Πάσκα. Το 2010 πρόεδρε είπαμε όχι στη συμφωνία TFTP όσον αφορά την χρηματοδότηση της χρητρομοκρατίας και την ενίχνευση των πηγών αυτής της χρηματοδότησης. Θέλουμε τώρα να γίνονται σεβαστά τα δεδομένα που αφορούν την ιδιωτική ζωή. Ε, έχουμε 80 εκατομμύρια τέτοια στοιχεία, φάκελους με στοιχεία. να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων με τη ΣΥΠΑ, με τρίτες χώρες, να υπάρχει αμοιβαιότητα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ισότητα όσον αφορά την ποιότητα και ποσότητα της πληροφορίας. Οπότε έχουμε εδώ κάποια προβληματάκια, το οποίο θα πρέπει να διορθωθούν όσον αφορά αυτή την συμφωνία που κατάλληλα είναι αξιόλογη. Όμως, θα πρέπει να δούμε ε, το τι θα γίνει με αυτό το είδος την, μαζική χίδιν ε, διαβίβαση δεδομένων. Κάτι το οποίο καταρχήν είναι Απαράδεκτο. Να υπάρχει λοιπόν χωρίς κανένα είδους ε, ε, ξεκαθάρισμα και ξεσκάρτωμα ε, μαζική διαβίωση δεδομένων. Επομένως θα πρέπει να, ε, ό,τι συμφωνείτε να είναι σύντονο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μόνο τα δεδομένα που έχουν σχέση με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και υπό τον διαβάζονται. Σε ευχαριστώ. Δύο λεπτά τώρα ο κύριος Κουέλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωτοσυμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με αυτή τη συμφωνία, είπα και ε. ε. Δηλαδή να υπάρχει εδώ πέρα κάποιο ε, δικαστική, αστυνομική αρρωγή βάση τη αμοιβαιότητα. Αυτό θα βοηθήσει όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια Είπαμε ότι κλείστηκε κάποια προσωρινή συμφωνία και τότε πριν των αρμοδιοτήτων είχαμε απορρίψει αυτή τη συμφωνία και τότε είχα πει τι αντιρρήσει μου, είχαμε πει ότι θα πρέπει πάντα η υπόψη προστασία των ε, δεδομένων. Τώρα, όμως το σκηνικό έχει αλλάξει. Υπάρχει συνεργασία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου Θέλουμε επομένω, επί τη βάση αυτών των αρχών, να διευκολυνθεί η μελλοντική συμφωνία μα με τη ΣΥΠΑ και να καταπολεμηθεί με επιτυχία η τρομοκρατία. Οπότε, έτσι λήφθη υπόψη το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 2009 και καλύφθηκαν αυτό το οποία θέλαμε, τόσο ώστε να υπάρχει αμοιβιότητα, να υπάρχει αναλογικότητα, Υπογραμμίζω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικές εγγυήσεις για μια ελάχιστη ε, περίοδο μετά την οποία θα πρέπει να διαγράφονται. Και θυμίζω την απέτηση για δυνατότητα ε, νομικής προσφυγής, επίσης ε, τον ορισμό καταλήλων εγγύσεων για την μεταφορά προσωπικών στοιχείων σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ελεγχθούν Και εκτό αυτού του πλαισίου δεν θα είναι δυνατόν να έχετε τη συγκατάβαση μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει στις αρχές που ανέκαθεν υπερασπιζόταν. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο και τώρα το λόγο έχει η κυρία Εμίν Μποσκούρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή ε, Κομισιόν, αγαπητό Συμβούλιο. Η πρότασή σας είναι ένα σωστό βήμα προς τη ε, σωστή κατεύθυνση η καταπολέμηση της τρομοκρατίας προέχει. Γι' αυτό θα πρέπει το συντομότερο να έχουμε μια νέα συμφωνία για τα SWIFT, αλλά όχι με κάθε τίμημα. Το Φεβρουάριο με μεγάλη πλειοψηφία απορρίψαμε μια κακή ε, ενδιάμεση μεταβατική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, το Κοινοβούλιο προσωπεί 500 εκατομμύρια πολιτών. Δεν θέλουν οι πολίτες τα τραπεζικά τους στοιχεία έτσι, χωρίς καμία εγγύηση να πηγαίνουν στις ΗΠΑ θέλουμε μια συμφωνία που να ε, εγγυάται και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε με την εντολή αυτή, τότε η κατάσταση διαφέρει σε πολύ μετά όσα έγιναν το Φεβρουάριο. Ε, ε, δώστε μας ένα λόγο για να μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε αυτή τη φορά. Θέλετε να ενημερώνετε το Κοινοβούλιο και καλά κάνετε που λαμβάνετε υπόψη σας καταγγελίες του Κοινοβουλίου και ε, για τις εγγύσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτά θα πρέπει να είναι τα κριτήρια και να υπάρχουν κριτήρια για το εάν θα πρέπει να διαβιβάζονται ή όχι τα στοιχεία ε, των πολιτών. Ε, και μόνο για την τρομοκρατία. Ωραία λόγια είναι όλα αυτά, ωραίες προθέσεις, αλλά θέλω να δω πώ μπορείτε να τα εγγυηθείτε στην πράξη. Η αρχή τη αναλογικότητα, τη αποτελεσματικότητα, προέχουν. Και η αμοιβαιότητα που είναι, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα έχουν την ίδια δράση. Αν δεν έχουμε μια ε, πλήρη εξήγηση και λεπτομερή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουν ε, να επιφορτιστεί ένας ε, ευρωπαϊκός οργανισμός με τον έλεγχο και την εξέταση των ετοιμάτων που θα έχουμε από τις ΗΠΑ. Πώς τη φαντάζεστε αυτή, Θέλει δικαστική αρχή. Οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα προσφυγής στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, σε δικαστή, ε, γιατί στην Ευρώπη έχουν αυτό το δικαίωμα. Παρακαλώ μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλεξάνδρ Άλβαρο. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε με επίση. Η εντολή που μας φέρετε τώρα δείχνει κυρίως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κυβούλιο είναι ξανά στην ίδια γραμμή. Είναι καλά αυτό που μας λέτε. Το Φεβρουάριο εμείς αρνηθήκαμε, απορρίψαμε τη συμφωνία. Ορισμένοι το θεώρησαν αυτό λεονταρισμό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με λεονταρισμό. Αυτό είναι αίσθημα ευθύνη. Ανάληψη ευθύνη για τα δικαιώματα εκείνων που εμεί εδώ εκπροσωπούμε, του Ευρωπαίου πολίτε. Οι τωρινέ διαπραγματεύσει για τη νέα συμφωνία θα πρέπει να απαντήσουν στο εξή κομβικό ερώτημα τι γίνεται με το σεβασμό, αγαπητό Κοινοβούλιο, τι γίνεται με το σεβασμό, αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέναντι ε, σε εταίρους, σεβασμό προς τους πολίτες και σεβασμό προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Νομίζω ότι στη νέα διαπραγματευτική εντολή έχουν μπει πολλά από εκείνα ε, που μας απασχολούσαν και τα θεωρούσαμε σημαντικά, καθώ επίσης και το ψήφισμα που θα εγκρίνουμε το Μάιο. Όλα τα μελήματά μας για την προστασία των πολιτών και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα δικαιώματά τους μπορούν με ετεροδικία να παραβιαστούν. Ε, έγινε μεγάλος λόγος για τις συλλογικές μεταβάσεις δεδομένων, ε, τα λεγόμενα bulk data. Τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει στη διαπραγματευτική εντολή τη τελική να ε, ορίζεται πώς και πότε θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να Υποστηρίζουμε αυτά που τώρα λέμε. Το ψήφισμά μας το αναφέρει αυτό σε δύο σημεία, διαπραγματευτική εντολή σε ένα και μόνο, αλλά νομίζω ότι θα βρει έναν τρόπο σοφό να το λύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. και παρακαλώ να κρατάτε το χρόνο σας. Ένα λεπτό έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο μέρες πριν να συναντηθούν οι υπουργοί των 27 κρατών μελών και να συζητήσουν το ίδιο θέμα γίνεται η συζήτησή μας. Ας είμαστε ειλικρινείς λοιπόν. Εμείς προσπαθούμε να ασκήσουμε πολιτική πίεση. Συζητούμε ένα πρόβλημα ενώ προσπαθούμε να σχηματίσουμε τη διαπραγματευτική εντολή για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Έχουμε μόνο δύο, δύο μήνες και μία ε, εβδομάδα μέχρι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει αυτές και η Κομισιόν εδώ δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτη με όλη την, ε, το σεβασμό στην Επίτροπο γιατί δεν ε, προτείνει καμιά εναλλακτική λύση. Άρα λοιπόν ε, τι μας λέει ή αυτό ή τίποτα αυτό είναι ενάντια στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν οδηγεί πουθενά, είναι αδιέξοδο. Φυσικά είμαι υπέρ της συνεργασίας, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δεν είμαι μεγάλος λάτρης του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά το θέμα είναι τι θα συμβεί αν η συμφωνία αυτή αντικρούσει τις θεμελιώδεις αξίες μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπάφτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι εντυπωσιακό για μένα που αυτή η Επιτροπή επιμένει να δίνει ελβέστητες οικονομικές πληροφορίες για εκατομμύρια πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ηνωμένου Βασιλείου παρά το, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών απέρριψε τις προτάσεις. Εδώ δεν είναι το θέμα πώς θα διαχειριστούμε μια συμφωνία SWIFT αλλά το να μην υπάρξει καθόλου SWIFT, συμφωνία SWIFT. Είμαστε κατά του χειρισμού και της παράδοσης στοιχείων στην Αμερική πολιτική. Αυτό μας οδηγεί σε έναν τρομακτικό μεγάλο αδελφό για την Ευρώπη. Σύμφωνα με τους, κανονικούς, με τους ισχύοντες κανόνες, 90 χρόνια μπορούν να διατηρούν τα στοιχεία η ΕΠΑ. Και αν και οι ΕΠΑ λένε ότι θα διαγράφουν τα στοιχεία μετά από 5 χρόνια, οι αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν ήδη κατηγορηθεί γιατί δίνουν τα στοιχεία σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείε όχι για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία, αλλά για να εξυπηρετήσουν οικονομικά συμφέροντα. Μια ενδιάμεση συμφωνία έχει ήδη υπογραφή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρί την κοινοβουλευτική συγκατάθεση. Γιατί η συνθήκη τη Λισαβόνα θα το είχε εμποδίσει αυτό, θα ήταν συναπόφαση. Και πάλι εμεί απορρίψαμε την ενδιάμεση συμφωνία και μία εβδομάδα πριν από αυτό η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών απέρριψε τη συμφωνία. Το, το εξακολουθείτε να συζητάτε αυτή την συμφωνία δείχνει την περιφρόνησή σα για τη δημοκρατία και για του λαού τη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ζουν στην δική μου περιφέρεια, την, στην Ουαλία. Η κυρία Μόνικα Χολμάγερ για δύο λεπτά. Äh, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αντίθεση με τον προλαλήσαντα, θα ήθελα να απευθυνθώ στην Επίτροπο Μάλσον και στην Επίτροπο Ρέντιν και να τις ευχαριστήσω για τις προσπάθειές τους εντατικές να ε, ανταποκριθούν στα μελήματα και στα προβλήματα που είχε θέσει το Κοινοβούλιο για τα προσωπικά δεδομένα, για το εμπιστευτικό ε, όλα αυτά τα λάβατε υπόψη για να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε. Επίσης, και άλλα ζητήματα που είπαν οι συνάδελφοι περιλαμβάνονται στη νέα εντολή. Τα έχετε σκεφτεί, τα έχετε επεξεργαστεί. Και εδώ αναφέρομαι κυρίως στην αμοιβαιότητα, στην αναλογικότητα και πάλι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχουμε τη δυνατότητα να ζητούμε ε, απάλληψη των ε, στοιχείων μετά από πέντε χρόνια να τα σβήνουν, να μην τα κρατούν για πάντα. Επίσης τα πρόστιμα. Όταν έχουμε ε, υπεξαίρεση των στοιχείων και χρησιμοποίησή τους για άλλους σκοπούς, να είναι απαγορευτικά τα πρόστιμα προς παραδειγματισμό. Κάτι άλλο όμως που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ε, ότι θα πρέπει να έχουμε ένα δικό μας TFTP ξεχωριστό και να μην ε, μεταβιβάζουμε μαζικά μεγάλους όγκους στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν έχει να κάνει με καχυποψία, καμία σχέση, αλλά με ισοτιμία και με ευθύνη και ακριβώς ε, να είναι στοχευμένη η παρέμβαση και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας με πραγματική ουσιαστική αμοιβαιότητα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κοιτάξει, ε, να το μελετήσει και να το συζητήσει με το, με το Συμβούλιο αυτό το θέμα του TFTP. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Τάνια Φαγιόν, Φαγιόν για δύο λεπτά. Η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τι βασικέ απειλέ στην ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χρειάζεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ για την ανταλλαγή οικονομικών στοιχείων όσο γίνεται πιο σύντομα, αλλά όχι με κάθε κόστο. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να προστατεύει του Ευρωπαίου πολίτε. Πρέπει να πετύχουμε μια καλύτερη συμφωνία που θα λάβει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και που θα λύσει το πρόβλημα των, των, της μαζικά ε, δεδομένων ε, η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Οι Αμερικανικές αρχές θα πρέπει επίσης ε, οι Αμερικανικές αρχές να μεταδίδουν ε, τα στοιχεία τους αν η Ευρώπη αποφασίσει να δημιουργήσει ένα δικό της πρόβλημα. Και είμαι ευτυχής που ακούω ότι η Κομισιόν συμφωνεί με το συγκεκριμένο σημείο. Είναι απαραίτητο να έχουμε καλές ασφαλιστικές δικλίδες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μέσω του οποίου το κάθε κράτος να μπορεί να εγκρίνει την μετάδοση, τη μεταφορά των ε, στοιχείων του. Και γι' αυτό και ρωτώ τι δυνατότητες θα έχουμε να απορρίψουμε τη, μεταφορά ε, προς τρίτες χώρες αν το αίτημα δεν είναι λογικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει TFTP, οπότε η ασφάλειά μας εξαρτάται από τις ΕΠΑ. Τι μπορούμε να αναμένουμε όμως σε αντάλλαγμα. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως ε, θα μπορέσουμε να <coughs> διακόψουμε τις συζητήσεις για τη συμφωνία αν δεν ανταποκριθούν στις δικές μας εγγύησεις στις δικές μας απαιτήσεις για εγγύησεις, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σετσίλια, Σεσίλια Βίκστρομ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μας ε, τους φιλελεύθερους από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ε, πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τις ε, διατελετικές σχέσεις ανάμεσα είπα, και Ευρώπη. Ε, όπως σε όλους τους τομείς. Αλλά επειδή σε όλους τους τομείς μπορεί να υπάρξουν περιπλοκές και δυσκολίες, θα πρέπει να επιλύονται. Ε, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν το να αντιμετωπίσουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Ε, κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, σαφές ότι πραγματικά ήταν ε, σκόπιμο το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέριψε αυτή τη συμφωνία. Όχι εδώ, εμείς εδώ στην αίθουσα θα πρέπει να καθοδηγούμαστε από την ε, δημοκρατία. Η συμφωνία η προηγούμενη για το SWIFT ήταν ελλειπής. Το Κοινοβούλιο ήδη εδώ και χρόνια είχε μιλήσει για τα δικά του τι δικέ του επιθυμίε. Τα κριτήρια περί του ψηφίσματος θα πρέπει να τηρηθούν και θα πρέπει από τη μια πλευρά να υπερασπιστούμε την ασφάλεια, αλλά από την άλλη πλευρά το δικαίωμα στην, στην ακαιρεότητα. Θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να δεσμευτούμε για αυτό το στόχο που είναι τόσο σημαντικός ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη αλλά και την ε, ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σιλβί Γκυγιώμα για δύο λεπτά. Όλοι θα συμφωνούσαμε όπως η καταπολέμηση τρομοκρατίας είναι κοινή ε, υπόθεση για την οποία, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει πλήρω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω είναι το ίδιο θεμελιώδη για εμά, του Ευρωβουλευτέ, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και ιδιαίτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων θα τηρηθεί. Είναι απαραίτητο να επιμείνουμε σε αυτό και αυτό δεν απευθύνεται μόνο ω μήνυμα στου εκπροσώπου τη Κομισιόν και του Συμβουλίου, αλλά και στι Αμερικανικέ αρχέ με τι οποίε θα πρέπει να διαπραγματευτούμε νέα συμφωνία. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα από πλευρά μου να υπογραμμίσω ένα σημείο το οποίο τονίζει τι βασικέ απαιτήσει συζητήσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Πρόκειται για το θέμα της διατήρησης των στοιχείων από τις Αμερικανικές Αρχές. Αυτό που προβλέπεται αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πως είναι δυσανάλογο και γι' αυτό και επιβάλλονται κάποια ερωτήματα. Για τι, ποιο λόγο να διατηρηθούν στοιχεία κατά τη διάρκεια πέντε ετών για στοιχεία τα οποία κατά τους συνομιλητές μας δεν θα χρησιμοποιηθούν. Δεν θα μπορούσε να μειωθεί αυτή η διατήρηση. Εν τω μεταξύ για τα στοιχεία τα πιο ε, που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν υπάρχει όριο. Ε, προηγουμένως προτινόταν τα 80 χρόνια, τα 90 χρόνια. Ε, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό να συνδεθεί με τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης έρευνας ή μιας συγκεκριμένης δίκης. Υπάρχει, προβλέπεται η χρήση αυτών των στοιχείων για άλλους στόχους εκτός της τρομοκρατίας και ποιοι είναι αυτοί. Μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά τα στοιχεία εδώ στην Ευρώπη και όχι στη ΣΥΠΑ. Θα ήθελα το Συμβούλιο και η Κομισιόν να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ενδώσει και είναι σημαντικό ότι το Συμβούλιο θα ε, υιοθετήσει την εντολή για την Κομισιόν να τα λάβει όλα αυτά ρητά υπόψη. Ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφε. Το λόγο έχει η κυρία Ναταλή Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ένα πολύ σημαντικό βήμα έχει γίνει πριν από δύο μήνε όταν αρνηθήκαμε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία. Χωρί να επανέλθουμε, γιατί η είμαι 27η ομιλήτρια απόψε για το ίδιο θέμα, θα ήθελα απλώ να τονίσω πω ορισμένοι ε, με ιδιαίτερο λυρισμό χαρακτήρισαν αυτή τη φάση τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία ω την πρώτη μέρα ύπαρξη του Ευρωκοινοβουλίου στο πλαίσιο τη Λισαβόνα. Όντω ήταν μια ιστορική σημασία νίκη, όχι μόνο λόγω του σεβασμού της ιδιωτική ζωή και της ελευθερία των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά ήταν και μια νίκη, ένα βήμα πολύ σπουδαίο για το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ ταυτόχρονα ήταν μια μεγάλη στιγμή θάρρους και παρησίας από πλευράς της δικής μας συζητήτης της κυρίας Χάνης Πλάσκα, την οποία θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα για... και μάλιστα σε μια στιγμή πολύ σημαντική για την ίδια. Θέλουμε να τονίσουμε την ανεξαρτησία μας, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, θα πρέπει ωστόσο να εξευρεθεί ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά και την ελευθερία των ανθρώπων, των πολιτών. Άρα λοιπόν αυτή η νέα εντολή θα πρέπει να μας καθοδηγήσει ώστε να βρεθεί μια δίκαιη, ισόρροπη ε, συμφωνία που θα σέβεται τους ε, νόμους ε, και καθώς και θα προστατεύει την ιδιωτική ζωή ώστε την προστασία δηλαδή των Ευρωπαίων πολιτών με λίγα λόγια, πράγμα το οποίο αποτελεί και τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, τα, για πολλούς από τους συμπολίτες μας και, και μου της ιδίας επίσης. Δεν επανέρχομαι στα θέματα αμοιβαιότητας, αυτά έχουν ήδη υποθεί, αλλά θα ήθελαν όλα αυτά να υποθούν με μεγάλη προσοχή και απαιτήσει ε, να μην δίνονται μαζικά στοιχεία πέρα από το δικαίωμα αποθήκευσης, το δικαίωμα τροποποίησης, το δικαίωμα ε, διαγραφής στοιχείων καθώς και το δικαίωμα νομικής προσφυγής. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσει ασφάλειας και τις απαιτήσει ελευθερίας. Ευχαριστώ. Grazie, Ευχαριστώ κυρία Γκρίσμπεκ. Σα συγχαίρω για την ακρίβειά σα. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Σένσιου για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε όλη τη σημασία που έχει παγκοσμίω η ανταλλαγή πληροφοριών στην καταπολέμηση τη τρομοκρατίας. Ε, η ομάδα μας υποστηρίζουμε κάθε δράση που ε, μπορεί να οδηγήσει στην ε, πάταξη της τρομοκρατίας εμείς εκπροσωπούμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε εκλεγμένοι βουλευτές. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους ε, υπερασπιζόμαστε γιατί υπάρχουν συνθήκες και συμβάσεις. Ε, ορισμένα πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η νομική προστασία, ε, η αμοιβαιότητα, η αναλογικότητα, τα εχέγγυα για την προστασία των δικαιωμάτων, η πάγια συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά τα θέματα. Ε, όλα αυτά ε, είναι πολύ σημαντικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εγγύησης ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι ε, τα στοιχεία αυτά είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία ε, των υπόπτων ή των πολιτών και να μπορούν οι πολίτες να προσφέγουν σε κάποια αρχή για να προσβάλλουν αυτές τις αποφάσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο και μετά από διαπραγμάτευση θα μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, ε, να προλάβουμε οποιαδήποτε παρατυπία, ατασταλία, να λύσουμε οποιαδήποτε ε, προβλήματα και σας ενημερώνω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και στις εθνικές αντιπροσωπίες έχουμε επαφές ε, με ε, τους ομολόγους μας και συνανόμαστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσάρς Γκέρνς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαλκυστίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου για το θέμα του SWIFT μπορεί να αποβεί σωτήρια υπό την έννοια ότι η συλλογή και η διαβίβαση των δεδομένων και των τραπεζικών στοιχείων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πολέμηση της δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω, είναι προφανές ότι ε, αυτό είναι πάρα πολύ αβέβαιο ένας ε, υποτιθέμενος, φερόμενος τρομοκράτης ε, που γνωρίζουν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι υπηρεσίε του δεν σημαίνει ότι είναι σημασμένο και στην Ευρώπη, όπως το δείχνει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτησή μου. Θα πρέπει να είναι στοχευμένη λοιπόν η συλλογή στοιχείων, να γίνεται με σεβασμό, με αμοιβαιότητα και εκεί θα πρέπει να βασιστεί οποιαδήποτε νέα συμφωνία. Νομίζω είναι σκόπιμο επίσης να σκεφτούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ε, να επιβάλλουμε το σεβασμό αυτών των ε, δικαιωμάτων και των ε, εξουσιών του Κοινοβουλίου. Και σε αυτό εναπόκειται να το πράξει. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριος Δερόσα. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζει τη συζήτηση αυτή και ε, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δέχτηκε πολλά από εκείνα που ζητούσε το Κοινοβούλιο όταν απέριψε την ε, αδόκιμη ενδιάμεση συμφωνία. Στις 6 Μαΐου θα ψηφίζουμε και καλό επιγόντως το Κοινοβούλιο να μην διεκπαιρεώσει καμία συμφωνία πριν την ημερομηνία αυτή. Η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου είναι απέτηση από τη συνθήκη και από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί έτσι ελαφρά την καρδία να συμφωνεί στο Συμβούλιο χωρίς να έχει δώσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Μικρή είναι η καθυστέρηση και θα είναι πολύ μικρή ε, η μικρότερη η ζημία στη σχέση μας με τις ΗΠΑ από μια δεύτερη απόρριψη από πλευράς Κοινοβουλίου χρειάζεται έλεγχος, ε, κοινοβουλευτικός έλεγχος. Μέχρι στιγμής δεν είμαι ικανοποιημένος από τα όσα μας προτείνονται. Εγώ θέλω πιο στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και στα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Ντερόσα. Και τώρα ακολουθεί η διαδικασία των αυθαρμήτων τοποθετήσεων Catch και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώ πως λέξη όπω είναι γνωστό, ο σκοπό αυτό είναι κοινό σκοπό και στόχο, δηλαδή η καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Αντιαμερικανισμό όμω ε, είναι κάτι που δεν το συμμεριζόμαστε όλοι. Να, ποια είναι η διαφορά επομένω μεταξύ ημών και των άλλων συναδέλφων των άλλων πολιτικών πτερίων. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να, να μπαίνουν τέτοια συναισθήματα μεταξύ ημών και του στόχου τη καταπολέμηση δηλαδή τη τρομοκρατία. Είναι κοινό εχθρό η τρομοκρατία. Επομένω, α κάτσουμε και να εκμεταλλευτούμε ό,τι δυνατότητε προσφέρονται τόσο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει επομένω η αμοιβαία εμπιστοσύνη μα να μην υπονομεύεται. Να, σε τι θα ωφελήσει το να προσυπογράψουμε και μεν και την συνθήκη SWIFT. Λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών κλπ. Όλα αυτά πρέπει να ε, τα, τα μολυμηθούν και επομένω με του συμμάχου μα από τη ΣΥΠΑ θα πρέπει να συμπορευτούμε. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Ζέιμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, Νομίζω ότι υπάρχουν ένα-δύο πραγματάκια τώρα τα οποία εδώ θα πρέπει να τα δούμε. Έχουμε εδώ πέρα την ε, Ατλαντική Συμμαχία, την εξωτερική πολιτική, την καταβλέψη τη τρομοκρατία, αλλά φυσικά και τη συνεργασία μα σε επίπεδο θεσμικών οργάνων για τη συνθήκη τη Λισαβόνα μα έχει προσδώσει νέε αρμοδιότητε, νέα, ε, νέα δικαιώματα. Οπότε μεταξύ των άλλων έχουμε τώρα και το θέμα τη προστασία των δεδομένων των συμπολιτών μα. Προστατεύσουν το θετικό του βίο, τη ζωή του. Επομένω, Γι' αυτό και θέλουμε μόνο όταν υπάρχει ε, στοχοθετημένη διαβίβαση δεδομένων να γίνεται να μην έχουμε υπερβολές σε αυτή τη ρύθμιση. Άρα εδώ να κάτσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Στη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και του στόχου μας. Μεταξύ αμοιβιότητας και αναλογικότητας και ασφάλειας των δεδομένων. Γι' αυτό σας λέω κύριε Υπουργέ, πού ήσασταν σήμερα το πρωί που θεωρούσαμε τα, του της κρίσης του 2008 γιατί για υπέρεπηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Δεν ήσασταν εδώ. Απουσιάζατε. Μέγαρα παρόλα ώρα. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπρόντς. One of the crucially important questions. Ένα από τα κρίσιμα ε, και πιο σημαντικά ερωτήματα είναι αν τα μαζικά στοιχεία θα πρέπει να μεταφέρονται ή αν θα πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα άτομα. Υπάρχει βέβαια και ενδιάμεση θέση. Οι ομάδες ε, πληθυσμού που συνδέονται με τρομοκρατία ε, θα μπορούσαν να στοχευθούν. Για παράδειγμα, αν ξαφνικά οι ψαράδες του Κόκνε άρχιζαν να σκοτώνουν ανθρώπους και όχι μόνο ψάρια, τότε θα πρέπει να στοχευθούν. Αν ηλικιωμένοι υπέρβαροι, συνταξιοδοτημένοι δάσκαλοι ε, γυμνασίου άρχισαν να σκοτώνουν τους μαθητές τους αντί να τους αναγκάζουν να πεθαίνουν από ανία μέσω των μαθημάτων που δίνουν τότε θα πρέπει να στοχευθούν ως ομάδα κάτι τέτοιο είναι κοινή λογική ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αποφυγή της μετάδοσης αυτών των στοιχείων που ανήκουν σε αθώα αθώους πολίτες. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόντζ. Το λόγο έχει η κυρία Ροϊτόβα. Πρόεδρε, ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι η ανάγκη εντοπισμού των χρηματοπιστωτικών ροών. Το Φεβρουάριο η αριστερά απέρριψε την ενδιάμεση συμφωνία χωρίς να προτείνει μια λύση και κατέστησε την ε, δουλειά της αστυνομία πολύ πιο δύσκολη. Θα πρέπει τώρα να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε μια νέα ε, μορφή συμφωνίας. Είμαι ευχαριστημένη που το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, είναι ανοιχτά, αλλά πραγματικά θα αφιβάλλω για το αν θα πρέπει να δίνονται όλα αυτά τα στοιχεία το κάθε μήνα. Μήπως θα υπάρχει δυνατότητα νομικής προσφυγής εάν υπάρχουν υποψίες και ποιος θα ελέγχει τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται στην Αμερικανική κυβέρνηση. Νομίζω πως θα πρέπει να υπάρχει μια μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή σύμφωνα με τι διεθνεί συμφωνίε και όχι η Ευρωπόλ γιατί η Ευρωπόλ δεν έχει αντίστοιχε αρμοδιότητε. Ή αλλιώ θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώ τη. Η δική μου προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατία. Δεν θα πρέπει να παρακάμψουμε τον, το χάρτη του θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να εγγυάται αυτά τα στοιχεία. Είναι απαραίτητο να δίνονται δυνατότητες προσφυγής σε περιπτώσεις αμφισβήτησης. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γιατεμάκη. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι ε, δεν ε, συμβάζονται πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σήμερα συζητούμε το SWIFT και βλέπουμε τι πρόβλημα έχουμε να διαφυλάξουμε τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών μας και να καταπολεμήσουμε ταυτόχρονα την τρομοκρατία. Βλέπουμε μεγάλα σύνολα δεδομένων να ε, διαβιβάζονται, να ε, αποθηκεύονται και να διατηρούνται για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η διμερή συμφωνία είναι χρονικά περιορισμένη, λίγη κάποτε και πότε σβήνουν αυτά τα στοιχεία στην πραγματικότητα από τη μνήμη. Ευχαριστώ. Μίλησε η κυρία Βέρτμαν βέβαια. Ε, θα σας δώσω, θα πήρατε μόνοι σας το λόγο, αλλά θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γιατεμάκη. η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι πολύ σημαντική και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετέχει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των ατομικών δικαιωμάτων. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι από τα πιο σημαντικές αξίες στην Ευρώπη και θα πρέπει να αποτελέσει και βασικό παράγοντα για την υπερδιατλαντική ε, συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει η διατλαντική συνεργασία και να λειτουργήσει αμφίδρομα. ανταλλαγή των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται για συγκεκριμένα άτομα και θα ήθελα επίσης να τονίσω πως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως ε, δικαιολογία για να καταπατήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως συνεργαζόμαστε με τους τρομοκράτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λόπες Γκαρίντο, κυρία Επίτροπε. Θέλω να συγχαρώ, σας συγχαρώ για την ε, ε, ε, νέα εντολή. Το ψήφισμά μας ε, συμπεριλαμβάνει τα, τις απαιτήσεις μας για την ασφάλεια αλλά και για την προστασία των δεδομένων και τον σεβασμό των θεμελιδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Το να οριστεί μια Ευρωπαϊκή Αρχή με νομικό χαρακτήρα ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με το, με το αντίστοιχο Υπουργείο των ΗΠΑ ε, νομίζω πως είναι πολύ καλή ιδέα. Είδα ε, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη μεταφορά μαζικών, ε, μαζική μεταφορά στοιχείων. Θα μπορούσαν και οι ευρωπαϊκές αρχές και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν στοιχεία για τις χρηματοπιστωτικές αναλλαγές που, συναλλαγές που αποθηκεύονται στη ΣΥΠΑ. Η συμφωνία SWIFT εξαρτάται από τις, τη σεβασμό των δημοκρατικών μας αρχών που πρέπει όλοι να εγγυηθούμε για χάρη των πολιτών μας. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε κυρία Νεντελτσέβα και τώρα φτάσαμε στην παρέμβαση του κυρίου Βαντερ Όχι, ναι, όχι, εντάξει. Σας ευχαριστώ. Τότε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λόπες Γαρίντο, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στα Ιταλικά ο υπουργό. Θα ήθελα καταρχάς να πω στον κύριο Σέμπερ ότι σήμερα το πρωί στη συζήτηση που αναφέρθηκε ήμουν παρόν. Ακόμα και αν δεν με είχαν καλέσει επίσημα, μου ζητήσατε να έρθω και ήρθα και μίλησα κιόλα και παρόν ήμουνα και απ' όλα. Μήπως εκείνος ήταν αυτός που απουσίαζε, όπως και τώρα απουσιάζει, γιατί βγήκε από την αίθουσα. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι η συζήτηση που κάναμε ε, σήμερα ε, μου φαίνεται άκρος επικοδομητική. Αντανακλά πραγματικά το πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει κατέρωθεν και ε, αυτό αφορά όλα τα μέρη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Χένις Πλάσχαρτ, ε, την συγκήτρια που μας το αναγνώρισε και την ευχαριστώ ε, για τη συνεργασία που είχε και με το Συμβούλιο και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ που το δηλώνει και δημοσίως. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η εντολή αυτή που πρότεινε η κυρία Μάλστρομ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και η εντολή που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα λάβουν υπόψη του τις ανησυχίες ε, του Κοινοβουλίου και θα εμπνευστούν από ε, τα δικά σας μελήματα και από το σχέδιο ψηφίσματος ε, της εισηγητρίας. Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που σας ανησυχούν και σας δυσκολεύουν, σας προβληματίζουν. Ε, οι ανησυχίες αυτές θα ληφθούν υπόψη στις κατευθυντήριες γραμμές ε, της διαπραγμάτευσης που θα εγκρίνει το Συμβούλιο. Η διαπραγμάτευση βεβαίως είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα καταλήξει ε, σε μια συμφωνία που θα υπογράψει και το Συμβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, κατευθυντήριες γραμμέ διαπραγμάτευσης. Το θέμα που επανειλημμένα ακούστηκε σήμερα. Η μαζική διαβίβαση δεδομένων, το είπε ο κύριος Άλμπρεχτ, Μπούσουτιλ, Σίπερ, η κυρία Σαρσεντίνη, Φένσον, Πάσκα, Ρόσα και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ε, βουλευτές ε, αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας πω ότι προφανώς και δεν μπορούμε να δεχτούμε αδιάκριτη μεταβίβαση στοιχείων, ό,τι και αν ζητούν και για οποιοδήποτε στόχο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Περί τίνος πρόκειται. Περί στοιχείων που μας ζητούν αποκλειστικά για την πρόληψη και τη διερεύνηση και τη δίωξη ε, αδικημάτων ε, τρομοκρατίας και χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Και μάλιστα με προσωποποιημένη στόχευση για πρόσωπα όπου έχουμε βάσιμες υποψίες ότι συνδέονται με την τρομοκρατία ή τη χρηματοδότηση αυτής δεν πρόκειται καθόλου για μαζική ε, μεταβίβαση στοιχείων. Όχι. Έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο και ένα υποκείμενο και αντικείμενο και υποκείμενο που περιορίζουν τη μεταβίβαση στοιχείων με κάθε σαφήνεια. Επιπλέον θα υπάρξει και ε, Ευρωπαϊκή Αρχή μέσω της οποίας θα ζητούν οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, τα στοιχεία αυτά και εκ των υστέρων θα υπάρχει και έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς λειτουργεί αυτή η συμφωνία, πώς ε, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά. Είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο λοιπόν που έχετε να απαντήσει στις ανησυχίες σας. Έγινε επίσης λόγος για τη διάρκεια αποθήκευσης και διατήρηση των στοιχείων αυτών. είναι περίπου μια πενταετία. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος χρόνος ε, με ε, μια στοιχειώδη αποτελεσματικότητα. Θα φροντίσουμε να είναι ε, το συντομότερο δυνατό διάστημα και ο χρόνος που θα επιβάλλεται από το στόχο και μόνο και καθόλου παραπάνω. Αλλιώς δεν θα είχε κανένα νόημα. Πάντα εργαζόμαστε προς ένα συγκεκριμένο στόχο και ένα συγκεκριμένο υποκείμενο. Το ίδιο ισχύει για το δικαίωμα πρόσβασης, ε, χρησιμοποίηση των στοιχείων, όπως είπε ο κύριος Κοέιο που έχει αποχωρήσει αυτή τη στιγμή, ε, ε, στάθηκε πολύ σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν για τη διαπραγμάτευση εγγράφονται στο πλαίσιο που μας πρότεινε η κυρία Μάλστρομ ότι αυτά τα δικαιώματα είναι εξασφαλισμένα, εγγυημένα, ε, πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση βεβαίως και θα πρέπει να είναι διασφαλισμένα ε, στη συμφωνία και εγγυημένα και οι αρχές της αναλογικότητας και της αμοιβαιότητας και στην τελική συμφωνία και στη διαπραγμάτευση προηγουμένω. Επίση, η δυνατότητα προσφυγή και διοικητική και δικαστική. Αδιακρίτω. Καμία διάκριση με βάση την εθνικότητα ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτό ε, θα είναι επίσης εξασφαλισμένο. Γιατί ε, η κυρία επιση εξασφαλισμενο γιατι η κυρια μποσκουρ ανέφερε και η κυρία Βερζιά. Και απόλυτη αμοιβαιότητα. από την προηγούμενη συζήτηση. Μας είχε απασχολήσει αυτό. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ε, της διαπραγμάτευσης και της εντολής που θα εγκρίνει το Συμβούλιο. Συμφωνούμε με τα όσα είπατε κι εσείς και με τα όσα προτείνει το σχέδιο ψηφίσματος κυρίας Χένης Πλάσχαρτ. Θα ήθελα να σας πω ότι το Συμβούλιο δεσμεύεται απολύτως να εγκρίνει εντολή που θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολίτων και θα εφαρμόζει με κάθε πίστη και θα σέβεται το γράμμα και το πνεύμα του ε, νόμου της ΕΣΔΑ, της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να προσυπογράψει και την ΕΣΔΑ τους ερχόμενους μήνες. Αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, και τώρα, δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Μάλμστρομ, λέει, η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Βουλευτέ, ναι. Όντω, πάρα πολύ επικοδοματική αυτή η συζήτηση. Και εμεί προσεκτικά σημειώσαμε όλα όσα είπατε. Το Συμβούλιο απάντησε ένα σωρό ερωτήσει που θέσατε. Αλλά να προσθέσω και εγώ δύο-τρία πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα έχουμε όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται στο μυαλό μα. Θα υπάρξει αναθεώρηση ενωσιακή ε, και αυτό μπορεί να γίνεται και σε τυχαία διαστήματα, μη τακτικά, ε, θεώρηση έλεγχο των δεδομένων, ούτω ώστε να βλέπουμε με, αυτό, αυτή τη δειγματοληψία ότι γίνεται ε, σεβαστή συμφωνία. Επίση, από την άλλη μεριά, όταν κάποιο φέρεται ότι χρηματοδοτεί η τρομοκράτη, επίση θα είναι αντικείμενο αυτή τη διαδικασία και θα έχουμε επομένω κάποια δικαστική αρχή που θα περιλαμβάνεται επίση πριν δοθούν κάποια ε, δεδομένα και θα, ε, θα, θα είναι συναρμόδια και η δική μα η κοινοτική αρχή. Επίση θα έχετε ε, προβασιμότητα κι εσεί. Να δούμε τώρα πώ ακριβώ θα γίνονται όλα αυτά. Αυτό είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορώ να πω πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά όπως είπε και το Συμβούλιο, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να διαπραγματεύσουμε. Να βρούμε δηλαδή μια λύση σε αυτό το θέμα και να δούμε πώ θα γίνουν οι διορθώσει, πώ θα γίνει η προβασιμότητα. Δεν θα έχουμε δεδομένα σε τρίτε χώρε. Θα έχουμε μόνο ε, πολύ συγκεκριμένα δεδομένα που θα δίνονται και όχι μαζική διαβίβαση και μόνο για κατανόηση τρομοκρατία. και μόνο οι εθνικές ε, αρχές θα επιλαμβάνονται του ελέγχου του σεβασμού της, ε, του, των αρχών προσθέσεων των δεδομένων θα πρέπει όσον αφορά τη μαζική διαβίβαση να έχουμε κάποιον που να φέρει το ότι είναι υπόπτως τρομοκράτης. Και μόνο τα ασφαλή δεδομένα θα διαβάζονται ένα κομμάτι τους, ε, ένα κλάσμα πολύ μικρό από αυτά τα δεδομένα. Οπότε εμείς θα δούμε, θα διερευνήσουμε το πώς μπορούμε να δούμε πώς θα λιγοστέψουν ακόμη περισσότερο αυτά τα οποία διαβάζονται. Αλλά έχουμε διατάξεις δεσμευτικές που περιορίζουν την προσβασιμότητα σε αυτά τα δεδομένα. Επίση, αν γίνει κάποια διαβίβαση δεδομένων και διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τα όσα έχουν συμφωνηθεί, θα διακόπτεται αμέσω στη διαφήμιση. Γι' αυτό σα λέω, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ότι μπορούμε για το SWIFT να είμαστε γρήγοροι ε, στο να κλείσουμε τη συμφωνία. Υπάρχει εδώ πέρα ένα, ένα, ένα χάσμα, ένα κενό, ένα παραθυράκι ασφάλεια. Θα πρέπει αυτό να το κλείσουμε. Αλλά νομίζω ότι πάρα πολλά ερωτηματικά απαντήθηκαν όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και όλα τα άλλα τα οποία είπατε. Δείξαν οι Αμερικανοί μια στάση πάρα πολύ ανοιχτή. Ε, είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μα και να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά όμως με φάνταστο τρόπο να απαντήσουμε σε όλε τι ε, απαντήσεις και επίσης από ό,τι ξέρω ε, μια ομάδα βουλευτών θα ταξιδέψει στην Αμερική και εκεί πέρα θα λυθούν κάποια θέματα. Τώρα παράλληλα με ε, αυτά τα ζητήματα ψάχνουμε να βρούμε αν θα υπάρχει ένα καινούργιο NTFP, να έχουμε δηλαδή μια καινούργια αρχή ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι μια καινούργια άλλη προβληματική και θα πρέπει να τη διερευνήσουμε στο βάθος. Αυτό δεν είναι για τις διαπραγματεύσεις. Είναι εσωτερικό δικό μας θέμα. Φυσικά και χρειάζεται αμοιβαιότητα, αλλά να το δούμε και αυτό. Η ΔΕ Κομισιόν πρόθυμα να υποβάλει προτάσεις αν το θέλουν τα κράτη-μέλη. Γιατί ξέρω ότι και εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο περιμένετε πώς και πώς να προχωρήσει αυτό το θέμα. Άρα έχουμε αυτή τη συζήτηση προβληματική που είναι παράλληλη. Αλλά παράλληλο είναι και το έργο της συναδέλφου μου της Αντιπροέδρου Βίβιαν Ρέντινγκ που έχει αρχίσει να φτιάχνει ένα σχέδιο εντολής για προστασία δεδομένων μακρόπνο για όλες τις συμφωνίες με την Αμερική. Γιατί και αυτό θα πρέπει να το δούμε στο όλο τοπίο. Τέλος έχουμε αυτό το ηφαίστειο στην Ισλανδία που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα για πολλούς παντού σε όλο τον κόσμο, προβλήματα στο να ταξιδέψει ο κόσμος. Άρα και εσείς Βέβαια καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε να ψηφίσετε, όμως σας βεβαίω, Α, εδώ με παρουσία ε, Προεδρία εγώ εδώ είμαι. Και οι συνεργάτε μα είδαμε το σχέδιο του κειμένου, λάβαμε υπόψη ότι είπατε, ακούσαμε τι είπαν οι τέσσερι πολιτικέ ομάδε και όλα αυτά θα τα πούμε και στου ε, υπουργού. Εάν δεν αναλυθεί απόφαση στο Συμβούλιο, θα χάσουμε δύο εβδομάδε διαπραγμάτευση. Γιατί όπω σα είπα, είναι θετικοί οι Αμερικανοί. Θέλουν να προχωρήσουμε, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο. Οι διαπραγματεύσει είναι δύσκολε. Χρειάζεται να έχουμε κάποιο χρονικό περιθώριο και Πρέπει αυτό να το κλείσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Αλλά να το κλείσουμε και όσο πιο καλά γίνεται. Και θέλουμε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ψηφίσει πριν τι διακοπέ. Να αποφασίσουμε. Για να αρχίσουν οι παραδείγματα όσο γίνεται πιο σύντομα. Καταλάβετε το παρακαλώ. Σα διαβεβαιώ. Και η Κομισιόν και η Συμβούλιο σα ακούσαν πάρα πολύ προσεκτικά. Και όπω το είπε και η Προεδρία, θα λάβουμε υπόψη αυτά το οποίο είπατε και θα τα πούμε αυτά την Παρασκευή στο Συμβούλιο των Υπουργών. Euh, Ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία, όπως θυμήσατε και εσείς, θα γίνει στη μήνυ σύνοδο του Μαΐου. Σύμφωνα με τη μέση διάταξη ακολουθούν δηλώσεις Συμβουλίου και τη Επιτροπή.